As everybody, the voting card. Έχετε όλοι τις ε, κάρτες ε, για την ψηφοφορία, την ηλεκτρονική. Inside the machine. Τα έχετε βάλει στη, ε, στην, στο μηχάνημα. And to wait just for one more minute. περιμένουμε κανένα λεπτό ακόμα. Κάποιοι λείπουν.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 ahora sí, yo creo que ya vamos a... Me pidieron dos minutos. Μου ζήτησε δύο λεπτά, καθυστέρησε για πάνω από δύο λεπτά, αλλά μέσα θα πρέπει να ξεκινήσουμε κάποια στιγμή. Τώρα θα σας πω σχετικά με τις ψηφοφορίες και την εξέλιξη τους. Καταρχήν να σας ε, ζητήσω να είστε πολύ προσεκτικοί. Είναι περίπλοκη η ψηφοφορία σε κάποια σημεία, διότι βασίζονται σε προηγούμενες ε, ψηφοφορίες κλπ. Έχουμε λίγο 300 σελίδες ε, ψηφοφοριών. Θα προχωρήσω γρήγορα, πρέπει να είστε προσεκτικοί. Εντάξει, αν κάποια στιγμή θα σταματήσουμε, θα σταματήσουμε, αλλά Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Παράκληση. Ενδιάμεσα, αν γινόταν να κάνουμε κάποιο μικρό διαλυματάκι μετά από μία ώρα, έτσι για να πάρουμε μια ανάσα, Ποιο θέλει να πάει στην τουαλέτα. Εγώ το ζητώ για τον εαυτό μου τουλάχιστον. Θα ήταν πολύ ε, καλό εκ μέρου σας. Ναι, εντάξει. Θα δούμε λοιπόν πώς θα προχωρήσει η τροπολογία αλλά σίγουρα θα το λάβουμε υπόψη. Πρέπει να είμαστε λοιπόν προσεκτικοί για να προχωρήσουμε και γρήγορα. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικός, αλλά θα πάει πολύ γρήγορα. Ανοίγει, κλείνει η ψηφοφορία, αποτέλεσμα και προχωρήσουμε. Διαφορετικά δεν θα τελειώσουμε τα αύριο. Ραούλου. θα ήθελα να ζητήσω πριν από την τελική ψηφοφορία, πριν από την τελική ψηφοφορία λοιπόν, να έχουμε κανένα δύο λεπτά στη διάθεσή μας για να αξιολογήσουμε τα αποτέλεσματα. Ποτέ ε, δεν έτυχε να με διακόψετε τόσες φορές ενώ μιλούσα. Εντάξει, εντάξει, συμφωνώ. Αρκεί να με διακόπτετε συνέχεια. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε γρήγορα. Καταρχήν ε, άρθρα, μετά το παράρτημα, μετά τα εκτιμώντας ε, και το ψήφισμα. Κάποια στιγμή θα κάνουμε και ένα διάλειμμα, σύντομο, για να πάει ο καθένας εκεί που πρέπει και πριν από το τέλος της θα διακόψουμε για 5-10 λεπτά, όπως κάναμε και σε άλλες ψηφοφορίες, σημαντικές και μακροσκελείς. Να πω όμως το εξή. οι ψηφοφορίες δεν είναι εύκολες και απλές σήμερα και έχουμε κάνει κάποιες παραχωρήσεις στις ομάδες και έχουμε και κάποιες ονομαστικές τις ψηφορίες σε συμβαστικές τροπολογίες. Αλλά αυτό δεν θα πρέπει να δημιουργήσει κάποιες, κάποια προβλήματα, το ζήτημα είναι τεχνικής φύσης ε, και θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εκ των προτέρων ευχαριστώ όλες και όλους για την συνεργασία τους και για το πνεύμα που θα θελήσουν να επιδείξουν κατά τη διάρκεια αυτών των ψηφοφοριών. Λοιπόν, εάν θέλετε κάποια διευκρίνηση, φυσικά θα σας τη δώσω. Πρέπει να είμαστε όμως πολύ προσεκτικοί και παρακαλώ τους παρισταμένους να παραμείνουν σιωπηροί αναφέρομαι σε συνεργάτες ε, και άλλους που συμμετέχουν στην συνεδρίαση. Περνάμε λοιπόν στον ε, ψηφοφορία την πρώτη Συμβασμό yeah. συμβασμός 1 αρχίζουμε τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται Τροπολογία 467 είναι. Υπέρ. Συγγνώμη, αρχή τη ψηφοφορία. Ε, έληξη ψηφοφορία. Δεκτή. Τροπολογία 469. Έναρξη ψηφοφορία. Πέρας. Τι συνέβη. Μικρόφωνο παρακαλώ, μικρόφωνο. Πηγαίνετε πάρα πολύ γρήγορα. Αν δεν μας δίνει η διερμηνία γρήγορα τον αριθμό, δεν μπορούμε να φτάσουμε στο, ε, στη σωστή σελίδα πριν κλείσετε την ψηφοφορία. Αν θέλετε μπορούμε να κάνουμε την ψηφοφορία στα αγγλικά. Αλλά ε, εντάξει, αυτό δεν έχει σημασία. Οι υπόλοιποι θα χρειαστεί να, ακούν άλλε γλώσσε, πάλι θα χρειαστεί να περιμένουν. 469 λοιπόν ήταν η τροπολογία, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορία. Δεκτή. Κοιτάξτε. Ζητώ και στου βουλευτές να προσέχουν. Ξέρετε ποια, ποια είναι η σειρά των τροπολογιών. Οπότε να παρακολουθείτε το έγγραφο και να ψηφίζεται αναλόγως, διότι αν ε, χάνουμε χρόνο τότε δεν θα προλάβουμε στον, στο πρωινό, μας χρειαστούν παραπάνω ώρες. Συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 2. Συμβαστική 2. Ψηφίζουμε. Πέραση ψηφορίας. Δεκτό. Συμβαστική 2, δεύτερο ακόμα τμήμα, υπέρ, ε, συγγνώμη, ψηφίσμα, Πέρας. Δεκτό. Προφορική τροπολογία για το τρίτο τμήμα, την... Ποιος αντιτίθεται, όχι, ε, ψηφίζουμε τροπολογία, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Τμήμα 4. Αρχίζουμε τη πέρα, Πέρας. Δεκτή. Τμήμα 5. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. Τμήμα 6. Ψηφίζουμε. Η ερωτήμα 6. Ψηφίζουμε πέρα, Απορρίπτεται. Τμήμα 7. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία στο τμήμα 8. Ενστάσεις όχι. Ψηφίζουμε. Ναι, ναι. Υπάρχει ένσταση για την προφορική τροπολογία. Άρα δεν υπάρχει με 8. με στο τμήμα 9. Ε, Προφορική τροπολογία. Υπάρχουν ε, αντιρρήσει. Ψηφίζουμε. Ποιος, ποιος αρνητίζεται, έχει ένσταση. Ψηφίζουμε. Τμήμα 9. Προφορική τροπολογία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τμήμα 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 4, 7, 1 τροπολογία. Συγγνώμη, 4, 7, 6. 4, 76. Ένταξη. Πέρας. Δεκτή. 475. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 477. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 478. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 4-7-9 ε, ψηφίζουμε πέρας απορρίπτεται 4-8-2 τροπολογία ας ψηφίσουμε συγγνώμη 4-86 4-86 ψηφίσουμε Πέρας. Τέσσερα, οκτώ, έξι. Ψηφίζουμε. Τέσσερα, ογδόντα, έξι. Αρχίζουμε την ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τέσσερα, 87 ψηφίζουμε πέρασε απορρίπτεται 488 ψηφίζουμε πέρασε Δεκτή. 4,90 ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. 492. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. 493. Πέρασε. Απορρίπτεται. 494. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. 495. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. 496. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. 498. Όχι, όχι, συγγνώμη. 517. 517. 5-17. Ψηφίζουμε. Ψήφισε να απαντήσω. Πέρασε. Απορρίπτεται. 5-19. Έναρξη. Πέρασε. απορρίπτεται. 5.23 ψηφίζουμε mm. πέρασε δεκτή συμβαστική 3 πρώτο τμήμα ψηφίζουμε πέρασε Κυρία Κύριε Φράγκα. Μικρόφωνο παρακαλούμε. Δεν θέλω να σας κουράσω, νομίζω ότι ο προσδιορισμός της ε, ε, αερασταθμικής αλίας για πορευθεί. Λοιπόν, θα πρέπει να ψηφίσουμε τον, ορισμό, τον εναλλακτικό ορισμό της ε, αερασταθμικής αλίας. No estoy Αναφέρομαι ε, στον προηγούμενο συμβασμό διότι απορρίφθηκε η χωριστή ψηφοφορία σχετικά με την εραστεχνική αλία. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να ψηφίσουμε την ε, εναλλακτική, τον ελεκτικό ορισμό της ε, αεραστανικής αλίας. That has been rejected. Okay. Uh, Vamos a ver, lo que vemos es que eh, la parte 1... Κοιτάξτε, το τμήμα 1 εγκρίθηκε. Δεν εγκρίνεται το υπόλοιπο τμήμα, ειδικά το 6 και το 7, τμήμα 7. Το τμήμα που εγκρίθηκε ήταν αυτό που ανταποκρίνεται στο 7, το small scale που αναφέρεται στα αγγλικά. Αυτή είναι λοιπόν που παραμένει ως έχει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 στη συμβιβαστική εν μέρη μόνο εγκρίθηκε. Επειδή λοιπόν δεν εγκρίναμε τα άλλα μέρη, πρέπει να τα ψηφίσουμε τώρα. Δεν μπορούμε να μην ψηφίσουμε τις τροπολογίες αυτές, γιατί η συμβιβαστική κατέπεσε. Και δεν μπορούμε να αφήσουμε όλες τις τροπολογίες, πρέπει να ψηφίσουμε με τίποτα, όχι. Ε, εκρίθηκε όλος ο συμβασμός που δεν εκρίθηκε ήταν οι επιμέρους τροπολογίες, τα split vote, οι ε, χωριστές ψηφοφορίες. Λοιπόν, είναι, είμαστε αναπόλυτα συνεπείς και πρέπει να περάσουμε στο άρθρο 5. Τι λέει και Παύλα. να επιβεβαιώσω αυτό που είπε ο σκιώδης εισηγητής, είχε απολύτως δίκιο. ¿Alguna otra intervención? Άλλο επιθυμεί να λέει το λόγο. Κύριε Ρωμέβα Να επιβεβαιώσω αυτό που έλεγε ο συνάδελφος ε, Μιλάνου. Και εγώ έτσι καταλαβαίνω το ζήτημα. Bueno, parece que uh, en relación con, con la... Το σε ό,τι φορά τον uh, συνδεσμό 1, αυτός είχε εγκριθεί και όλα όσα περιλαμβάνει. Το τμήμα του συνδεσμού για το οποίο δεν υπερσφίστηκε, φυσικά απορρίφθηκε από πλευρά Κομισιόν της Επιτροπής, αλλά το τμήμα του ορισμού που μας ενδιαφέρει έγινε δεκτό. Δεν ξέρω τώρα πρέπει να περάσουμε στο που ήμασταν. Τροπολογία 524. 524 τροπολογία. Ψηφίζουμε. Έληξε ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Ψηφίσαμε λοιπόν τον σειρασμό 3 πρώτο τμήμα και τώρα περνάμε στο δεύτερο τμήμα του συμβασμού 3. Έναξη ψηφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. Πεντακόσια εξήντα δύο. 562 τροπολογία Ψηφίζουμε. Πέρας. Όχι, όχι. Έναρξη της ψηφορίας. Τι είναι, το δουλεύει το μηχανάκι σας. Εντάξει. Ξαναρχίζουμε. Έναρξη ψηφορίας. Πέρας. Ψηφίζουμε την 562. Δεκτή. Συμβαστική 4. Πρώτο τμήμα της Συμβαστικής Τροπολογίας 4. Έναρξη. Πέρας. Δεκτή. Δεύτερο τμήμα του συμβαστική τέσσερα έναρξη. Πέρασε. Δεκτή. Τρίτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Δεκτή. τέταρτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Δεκτή. Πέμπτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 582. 582. Ψηφίζουμε. Πέρας. Από την αρχή. 582. Ψηφίζουμε.

Πέρας. Απορρίπτεται. 608. 608. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 617. 617. Ψηφίζουμε. Πέρας. απορρίπτεται. 6.34 ψηφίζουμε πέρας απορρίπτεται 6.44 ψηφίζουμε πέρας απορρίπτεται 661. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 670. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 705. 705 στο άρθρο 7. Συνεχίζετε μπροστά σα. 705. Στο άρθρο 7. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 5. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Δεκτή. 710. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 53. τρία της Επιτροπής Απασχόλησης. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 6. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική 7 ψηφίσουμε. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 720. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική 8. Πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Ε, συγγνώμη, ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Τέταρτο τμήμα. Απορρίπτεται. Το επόμενο καταπίπτει το τμήμα 5. δεκτή. Τμήμα 6 ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτό. Τμήμα 7 ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτό. Εφτά πενήντα τέσσερα. Τροπολογία. 754 στο άρθρο 12α νέο. Το βρήκατε. Α, ψηφίζουμε. Όχι. Τι γίνεται, Μάικλ. Δεν λειτουργεί. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική εννέα. Έχουμε έξι τμήματα. Πρώτο το τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτό. Τρίτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτό. Τέταρτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Α, συγγνώμη, συγγνώμη, δεκτό, δεκτό, δεκτό. Σε περίπτωση ισοψηφία, όταν υπάρχουν χωριστέ ψηφοφορίε, ε, γίνεται δεκτό. Το επόμενο τμήμα 5, ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτό. Έκτο τμήμα. Ξεκινάμε την πληροφορία, Πέρας. Δεκτό. 758. 758. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτό. 759. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτό. 7-7-4. Ψηφίζουμε. Πέρασε Απορρίπτεται. 803. 803 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 807 ψηφίζουμε. Πέρας. απορρίπτεται. Συμβαστική 10. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτό. 814. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται 818. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτό. Δεκτή μάλλον τροπολογία. 820. Ψηφίζουμε. 820. Πέρα ψηφορίας. Δεκτή. 842. 842. 842 Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 11. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 19. Ψηφίζουμε. Τροπολογία 19 του προπολογισμού. Επιτροπής προπολογισμού. Το άρθρο 6α νέο. Ψηφίσατε. Πέρας ψηφορίας Δεκτή. Συμβαστική 12. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 863. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 13. Υπάρχει μια προφορική τροπολογία της κυρίας Τόμας. Ε, δώσω το λόγο πρώτο να περάσουμε. Α, την έχουμε την τροπολογία. Θα την αναγνώσω εγώ. Α, δύο μέλη ε, έχουν ε, αντίθετη γνώμη, άρα δεν ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε τώρα την συμβαστική 13. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 877. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 14. Σε τρία τμήματα. Όχι τέσσερα, τέσσερα τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεύτερο τμήμα. Το πρώτο έγινε δεκτό. Προφορική τροπολογία Υπάρχουν ε, συνάδελφοι που διαφωνούν, άρα δεν υπάρχει προφορική τροπολογία. Περνάμε στο τμήμα 3. Ε, ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Τμήμα 4. Ψηφίζουμε. Πέρας. Πέρα της Δεκτή. 880 τροπολογία. 880. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 881. Ψηφίζουμε. Πέρας της Δεκτή. 884. Ψηφίζουμε όπως και ταυτόχρονα με την 8 το 6 ψηφίσουμε ομού. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 8, 8, Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική 15 σε τέσσερα τμήματα κύριος Καντέκ. Μια μικρή παρατήρηση για να πω ότι υπάρχει μια μικρή αλλαγή στον κατάλογο ψηφοφορίας του ΕΛΚ σε σχέση με τα τμήματα 2 και 3. Είναι συν το πρόσημο, θετικό και όχι αρνητικό. Συνεχίζουμε πρώτο τμήμα της τροπολογίας της συμβιβαστικής πρωτοπολογίας 15. Ψηφίζουμε. <clears throat> Πέρασε. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα. Ξεκινάει η τροπολογική ψηφορία. Πέρας. Δεκτό. Τρίτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτό. Τέταρτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Α, υπάρχει προφορική τροπολογία. Υπάρχουν ε, αντίθετε γνώμε. Εντάξει, δεν την ψηφίζουμε τότε. Περνάμε στην 904, 904 της Ζαμπέλ Τομά. Ψηφίζουμε. Πέρα της ψηφορίες Απορρίπτεται. 949, 949 τροπολογία το άρθρο 21. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. Ένβη. Όχι, όχι. Συγγνώμη. Συμβαστική 16. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική 17. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτό. Τώρα περνάμε στον συνδυασμό 18. Ψηφίζουμε. Πέρας. Με το 19 και Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτός. Ο συμβασμός 19. Και τώρα περνάμε στο 9, Ευρωπαϊκή 979, στο άρθρο 26. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 9.80. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 20. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτό. Συμβαστική τροπολογία 21 σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτό. Τρίτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτό. Συμβαστική 22. Ψηφίζουμε. Απρίνα πριν από το Συμβασμό 22 την τροπολογία 1001. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. Και τώρα περνάμε στο συμβαστική 22. Ψηφίζουμε. Πέρας της ψηφοφορίας. Δεκτός. Συμβαστική 23. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτός. Συμβαστική 24. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 25 συμβαστική. Συμβαστική 25. εχει 4 4-5 τμήματα. Πόσα είναι. Πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτό. Το πρώτο τμήμα. Δεύτερο ναι. τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτό. Τρίτο τμήμα. Υπάρχει προφορική τροπολογία. Κάποιοι ενίστανται. Όχι. Ψηφίζουμε το τρίτο με την προφορική τροπολογία. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτό. Τέταρτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτό. Και... Και τώρα Περνάμε στο 1104, 1104. Το βρήκατε. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται η 1104. 11.09. Ψηφίζουμε. Πέρας. απορρίπτεται. 1110 ψηφίζουμε πέρας απορρίπτεται. Χίλια Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 1151. Ψηφίζουμε. Πέρας. 1151. Ψηφίσατε. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβασμός 26. Σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτό. Τρίτο τμήμα. Υπάρχει μια προφορική τροπολογία. Υπάρχουν ενστάσεις. Ναι, αλλά δεν υπάρχει. Περνάμε στον συμβαστική 27. Πόσα τμήματα έχει εδώ, από 8. Πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε. Ναι. Πέρας.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 Τέταρτο τμήμα. Μία ανακοίνωση. Από εδώ και στο δεν θα υπάρξει διερμηνία προς τα πολωνικά. Και υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Δεν θα έχουμε πολωνική διερμηνία. Τέταρτο τμήμα. Προφορική τροπολογία. Υπάρχουν ενστάσεις. Όχι. Άρα ψηφίζουμε την προφορική τροπολογία στο 64. Πέρασε ο φορείς. <coughs> Δεκτή. Τέταρτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Α, μισό λεπτό. Έκτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Δεκτό. Εβδο, τμήμα 7. Προφορική τροπολογία στο τμήμα οράλ. Υπάρχουν ενστάσεις, όχι, άρα ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτό. Και το τμήμα 8. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτό. Συμβαστική 28. Ψηφίζουμε. Πέρας δεκτός 1171 1171 ψηφίζουμε πέρας δεκτή συμβαστική 29 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα ψηφίζουμε πρώτο τμήμα λοιπόν στο 29 πέρας δεκτή Δεύτερο τμήμα, προφορική τροπολογία, υπάρχουν στάσει. Όχι. Δεύτερο τμήμα, το συμβαστική 29. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Και τώρα έχουμε τον συμβαστική 30. Συνεπιστική τροπολογία υπερθυμού 30. Άρθρο 33 Β νέο. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε άπαντες. Πέρας. Εγκρίθηκε. Προφορική τροπολογία παριθμών 6 της Άλντε. Υπάρχουν ενστάσεις. Ναι, άρα δεν τη ψηφίζουμε. Περνάμε στην τροπολογία. 101. Τροπολογία 101 μαζί με την 1199 ψηφίζουμε και την τροπολογία του προπολογισμού 22. 101, 1199 και του προπολογισμού 22. Στο άρθρο 34 ψηφίζουμε. Πέρασε. Δεκτή. Δεκτές μάλλον. 12.08.1208 ψηφίζουμε. Συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Περνάμε στην βασική κάνουμε ένα άλμα λοιπόν και φτάνουμε μέχρι την συμβιβαστική την επόμενη που είναι 31. 31, que se 31. Σε τρία τμήματα. Πρώτο Πέρας. Δεκτή. Δεύτερο βήμα. Δεκτό. Τρίτο τμήμα. Συγγνώμη, υπάρχει προφορική τροπολογία, υπάρχουν ενστάσει. Περνάμε στο επόμενο σημείο. Υπήρχαν τελικά ενστάσει. Περνάμε στην ευαστική 32. Και εδώ σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Δεκτό. Ε, συγγνώμη, έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεχτώ. Τρίτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεχτώ. Περνάμε στην 1288. 1288. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Δεκτή 1290. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. Ρέτζι 79. Άρθρο 36. Ένα νέο. Ψηφίζουμε. Πέρας. 79. Τροπολογία 79. Πέρας δεκτή. Τροπολογία, ε, συμβαστική 33 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτό. Τρίτο τμήμα καταπίπτει 3, 1317 ε, ψηφίζουμε πέρας απορρίπτεται συμβαστική 34 σε τρία τμήματα πρώτο τμήμα ψηφίζουμε πέρας δεύτερο τμήμα Ψηφίζουμε. Πέρα. Δεκτό. Τρίτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτό. Συμβαστική 35 σε πέντε τμήματα. Πρώτο τμήμα. Πέρας. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτό. Τρίτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτό. Τέταρτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτό. Και πέμπτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας απορρίπτεται το πέμπτο τμήμα 1382 1382 ψηφίζουμε πέρας δεκτό δεκτή 1384 ψηφίζουμε πέρας δεκτή 1385 ψηφίζουμε Πέρας. Δεκτή. Συμβεστική 36. Σφίζουμε. Πέρας. Δεκτός. 1423. 1423. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 37 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Πέρας. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε πέρας δεκτό και το δεύτερο τμήμα της 37 1472 ψηφίζουμε 1472 1462 1462 1462, όχι 72, 62. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 1478. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική 38. Σε πέντε τμήματα. Έξι τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα. Πέρας. Δεκτό. Τρίτο τμήμα. Πέρας. Δεκτό. Τέταρτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. λεκτό. Πέμπτο τμήμα υπάρχει προφορική τροπολογία. Υπάρχουν ενστάσεις. Όχι. Ψηφίζουμε το πέμπτο τμήμα λοιπόν της προφορικής τροπολογίας. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Υπάρχει και εδώ προφορική τροπολογία. Υπάρχουν στάσει Όχι. Ψηφίζουμε την προφορική τροπολογία. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. a Envi 122. Πάμε στην Envi 522. Σε ποια σελίδα, ρωτάει ο κύριος Καντέκ. Εμβι 122. Έναξη ψηφοφορίας. περασε απορριπτεται Απορρίπτεται. 15-15. Έναρξη ψηφοφορία. 15-15 και 15-16. Έναρξη ψηφοφορία. 15, 15, 15, 16 που είναι ταυτόσιμες. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. 15-17. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμπεβαστική 39. Πέντε τμήματα. Πρώτο τμήμα έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. τμήμα ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Πέμπτο τμήμα. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην 1535. 1535. Άννα Μιράντα. Έναρξη ψηφοφορίας. 1535. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 40, έναρξη. Δύο τμήματα, συγγνώμη. Πρώτο τμήμα. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα, έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 1552. Φερέιρα, έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. 1558. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. 1559. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 41. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, με προφορική τροπολογία της, κυρία Τόμας, της κυρίας Τόμας. Διαφωνεί κανείς? Δεν διαφωνεί κανείς, οπότε ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα με την προφορική τροπολογία της κυρίας Τόμας. Έναρξη ψηφοφορίας. παράγραφος 1 να προσθέσουμε offshore ε, mine plants. Edible mining plants. Αυτό προστίθεται. Λοιπόν, ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα με την προφορική τροπολογία. Διαφωνούμε, λέει ο κύριος ε, Ραούλη Ραμουέβα. Σηκώστε το χέρι παρακαλώ όσοι διαφωνείτε. Ωραία. Δεν ψηφίζουμε την προφορική τροπολογία. Το δεύτερο τμήμα χωρίς την προφορική τροπολογία. Όσο έχει το δεύτερο τμήμα. Έναρξη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 1583. Σάντσες Πρεσέδο. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 42. Έναρξη ψηφοφορίας. Συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος, έχει τρία τμήματα η συμβιβαστική 42. Πρώτο τμήμα. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Τρίτο τμήμα, το 2α κατέπεσε. Τρίτο τμήμα λοιπόν, έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. 16-20 τώρα. 1620. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 43. Τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται τρίτο τμήμα καταπίπτει, γιατί ψηφίστηκε το προηγούμενο. Συμβαστική 44. Δύο τμήματα, πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Πέτσου, 16.35. 16.35 τώρα. 16.35. Πρέπει να το ψηφίσουμε. Έναρξη ψηφοφορίας. Τόμας. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 44. Δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα το ψηφίσαμε. Πάμε στο δεύτερο τμήμα. Ε, μα το ψηφίσαμε και προηγουμένως αυτό. Το δεύτερο τμήμα της συμβιβαστικής 44 πρέπει να ψηφίσουμε τώρα. Συμβιβαστική 45. Απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα τότε. Τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα, έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα, έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται τρίτο τμήμα, έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται 1678. Δύο τμήματα. Αλλά ψηφίζουμε μόνο το πρώτο τμήμα, το non-legal. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 46 τώρα. Δύο τμήματα και πάλι. Πρώτο τμήμα, έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 46. Έναρξη ψηφοφορία. Συγγνώμη, 47. Έναρξη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 48. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 17-22. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 17-26. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 49. Πέντε τμήματα. Πρώτο τμήμα. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται τέταρτο τμήμα, έναρξη. Συγγνώμη, υπάρχει προφορική τροπολογία. Διαφωνεί κανείς? Όχι. Οπότε ψηφίζουμε το, ψηφίζουμε το τέταρτο τμήμα. Έναρξη ψηφοφορίας, πέρας. Απορρίπτεται. Πάμε στο πέμπτο τμήμα, έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 50. Τέσσερα τμήματα. Πρώτο τμήμα. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Όλο, όλη η συμβιβαστική καταπίπτει τότε. 1754. 1754. Ψηφίζουμε τώρα. Why? Θέλετε να ξαναψηφίσουμε γιατί. Δεν πρόλαβα να ψηφίσω. Ε, αφού είναι ηλεκτρονική η ψηφοφορία. Ε, ελέγχουμε όταν είναι με τα χέρια ψηφοφορία, αλλά άμα είναι ηλεκτρονική ψηφοφορία, άμα δεν σας αρέσει η ψηφοφορία, ξαναψηφίζουμε. Είναι Κύριε Μιλάνε, είναι ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρα δεν πρέπει να ελέγξω τίποτα, δεν πρέπει να κάνω κανένα τσεκ. Ε, κάποιος ή έχει ψηφίσει ε, ή μπορεί να μην έχει ψηφίσει, να έχει ξεχαστεί, να έχει αφαιρεθεί κλπ. Η ψηφίσει ε, ε, ναι ή όχι ή ε, ψηφίζει Πρόεδρε 200 ψηφοφορίες κάναμε και δεν ζήτησα κανέναν έλεγχο το μηχάνημά μου δεν λειτουργήσε γι' αυτό ζητώ να επαναληφθεί η τροπολογία αυτό είναι όλο Κοιτάξτε, εντάξει, μου ζήσατε έναν έλεγχο, ένα τσεκ, αλλά το μηχάνημά σας δεν λειτουργήσε, μια ψηφοφορία, μου το είπατε, και αυτό το οποίο δεν έχει έννοια κατ' είναι ότι να γίνεται έτοιμα για τσεκ όταν έχει βγει ήδη το αποτέλεσμα. Όταν είναι γνωστό το αποτέλεσμα. Γι' αυτό λοιπόν εκεί είναι η ένστασή μου. Ανάμεσα στο 524. 1754. Ψηφίσατε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Να μου το πείτε, αν δεν δουλεύει. Πρόεδρε, και εμένα μερικές φορές ε, δεν ε, μου λειτουργήσε το μηχάνημα, γι' αυτό θα πρέπει να υπολοιθεί γραπτός ε, το γεγονό ότι ψήφισα και ότι δεν ε, επηρέασε αυτό το αποτέλεσμα εμπέστος επειδή πηγαίνουν τόσο γρήγορα πρόεδρε μερικές φορές έτυχε να μην καταφέρουν να ψηφίσω εντάξει δεν υπάρχει πρόβλημα εντάξει το καταγράψαμε ευχαριστώ εν πάση περιπτώσει μπορούμε πάντα να προχωρήσουμε μόνο ότι το μηχανάκι πότε πότε κάνει και τα δικά του 17.55 έναρξη πέρας Απορρίπτεται. 1756. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. 1756 ψηφίζουμε τώρα. Απορρίπτεται. 1757. Έναρξη ψηφοφορίας. Ψηφίσατε. Πέρας. Απορρίπτεται. 1761. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. 1759. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. 1762 ψηφίζουμε τώρα. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. 1765. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 51, δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 52. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. 1797. 1797 έναρξη ψηφοφορίας. Ψηφίσατε. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 53. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. 18-16 και 18-17 που είναι ταυτόσημες. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας απορρίπτονται. 18-18 έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. 18-19. Α, καταπίπτει, καταπίπτει γιατί ψηφίσαμε την προηγούμενη, υπερψηφίσαμε την προηγούμενη. 18-20. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 54 τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Α, έχει καταπίπτει γιατί ψηφίσαμε το δεύτερο τμήμα και πέρασε. Συμβιβαστική 55 έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 56. Τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα έναξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα. Πρώτο τμήμα. Ε, συγγνώμη, έναρξη ψηφοφορίας. εγκρίνεται, το δεύτερο κομμάτι, το B, καταπίπτει. 18.59 τώρα. Μαρία Πατράου. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. 18.71. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας απορρίπτεται. 18.70 έναρξη πέρας απορρίπτεται. Περνάμε τώρα εμπλέο 78. Έναρξη ψηφοφορίας πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 57 έναρξη, πέρας, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 58, έναρξη, πέρας, εγκρίνεται. 1887, έναρξη, πέρας, απορρίπτεται. 1888 και 1889. Ταυτόσημες. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεκαοκτώ ενενήντα οκτώ. Δεκαοκτώ ενενήντα οκτώ. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Okay. 19.00. 19.00. 1900. «1901» ψηφίζουμε. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. 1902 έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. 1903 και 1904 έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας, εγκρίνεται. 1905 έναρξη ψηφοφορίας. πέρας, εγκρίνεται. 1906 έναρξη. Α, συγγνώμη. Καταπίπτει. 1908 τώρα. Ούτε. Ναι. 1907. ψηφίζουμε, έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. 1908. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. 1909. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική... Συμβιβαστική 59. Πήγα πολύ γρήγορα, δεν έχουμε φτάσει στην 60 ακόμα. Συμβιβαστική 59, έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. 19-14 ψηφίζουμε τώρα. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 60. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Ρέτζι 114. Άρθρο 70α, έναξη ψηφοφορίας. Ψηφίσατε. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 61 σε 5 τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Δεκτό. Τρίτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Δεκτό. Τρίτο. Α, έχει καταπέσει. Τέταρτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτό. Και καταπέφτει το 4α. Συμβαστική 72. Σε 62. 62. Σε δύο τμήματα. Ο συμβασμός είναι 62 το άρθρο είναι το 72. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτό. 1998 τροπολογία. Ψηφίζουμε. 1998. πέρας, Δεκτή. Ρέγγι 132. Ψηφίζουμε. Πέρα ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 2051. Ψηφίζουμε πέρας απορρίπτεται συμβασμός 63 με τέσσερα τμήματα πρώτο τμήμα πέρας δεκτό δεύτερο τμήμα ψηφίζουμε πέρας δεκτό τρίτο τμήμα ψηφίζουμε Τρία πρώτα τμήμα ψηφίζουμε. Δεκτό. Άρα το 3α καταπίπτει. Τμήμα 4 ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτό. Περνάμε στην ρέτζη 136. 136 ψηφίζουμε. Πέρας δεκτό. Συμβαστική 74. 64, συγγνώμη, ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτό. Συμβαστική 65, ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτός. Συμβαστική τροπολογία 66, ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική 67 σε δύο τμήματα. Συνδεπτά. Πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτό. 2093. 2093 του Τόμας. Της Τόμας μάλλον. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συνεβαστική 68. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτός. 21-11. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 21-12. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 21-21. Ψηφίζουμε. Πέρας απορρίπτεται 21-22 ψηφίζουμε πέρας απορρίπτεται 21-23 ψηφίζουμε πέρας δεκτή 21-26 21-26 ψηφίζουμε. Δεν υπάρχει. Πέρασε. Απορρίπτεται. 21-28. Πέρας. Απορρίπτεται. 21-33. 21-33. Πέρασε. απορρίπτεται. Συμβαστική 69 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Πέρας. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτό. Συμβαστική 69, ε, συγγνώμη, 70. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική. 71 σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτό. Τρίτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας δεκτό. 21, και NV 165 που είναι ταυτόσιμες. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτές. 72 τρόπο συμβαστική. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτός. Δεκτή. Ε, 2186 ψηφίζουμε. Πέρας, δεκτή. Η ένδυ καταπτύπτει. 2187. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική 73. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. Τρίτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Και τώρα 2196 τροπολογία. 21-146. 146. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 2197 Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 2198. Ψηφίζουμε πέρας δεκτή. 2199. Ψηφίζουμε πέρας δεκτή. 2200. Ψηφίζουμε πέρας απορρίπτεται. ΕΜΠΛΟ 84. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 22-01. 2-201. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 22-02. 2.202 ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. Συμβαστική 84. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ψηφίζουμε. Πέρας. Δεύτερο τμήμα. Πέρασε δεκτό. δεκτώ. 22-16, ψηφίζουμε. Πέραν δικτυακή. Συμβαστική 75 ψηφίζουμε. Έρα δικτύ. 22-26. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 22-41. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 22-72. κάνουμε ένα μεγάλο άλμα για το 2272 σελίδα 220 άρθρο 96 Τι βρήκατε? 2.272, 73 και 74. Είναι ταυτοσιμες Εντάξει. Ψηφίσμα. ψηφίσατε άπαντες πέρας απορρίπτεται 2246 2246 ψηφίζουμε πέρας απορρίπτεται 2271 ψηφίζουμε πέρας 2.275 Παναλαμβάνω 2.275 που είναι ταυτόσιμο με τη Ρέτζη 141 Είναι σε αυτές οι δύο Πέρα ψηφοφορίας Απορρίπτεται 2.276 ψηφίζουμε πέρας απορρίπτεται. 2.277 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 2.280 που είναι η αυτή με την 73 της ένδυ. Υπέρ, ε, συγγνώμη, ψηφίζουμε. Πέρας, απορρίπτεται. 2.272 και 2.273 είναι ταυτόσιμες ε, πέρας απορρίπτεται 22.44 ψηφίζουμε πέρας απορρίπτεται 142 ρέτζι ψηφίζουμε πέρας απορρίπτεται 22.85 ψηφίζουμε πέρας Απορρίπτεται. 2286. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. 2284. 2284 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Ένδυ 144 ψηφίζουμε. Πέρας απορρίπτεται. 22.87 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 22.88 ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 23.05 ψηφίζουμε πέρας μπορείτε 23, 06, 07, 08, 09, 010 που είναι ψηφίζουμε πέρας απορρίπτεται απορρίπτονται 48 ψηφίζουμε πέρας απορρίπτεται 2450 ψηφίζουμε πέρας απορρίπτεται 2347 ψηφίζουμε πέρας δεκτή κατέπεσε 2246 περνάμε στην 101 προφορική. Υπάρχουν ενστάσει. Ε, άρα δεν ψηφίζουμε, περνάμε στην τροπολογία 2451. Ψηφίζουμε. Πέρας. Έχεις δει το λόγο πριν από την ψηφορία. Όχι, αργότερα. 2451. Απορρίπτεται. 23.50. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Προφορική 8. Υπάρχουν στάσει Περνάμε στην 24.52. 24.52. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 24.53. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 24.54. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 24.51. 23.50 Και 176. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 23, 52, έχει καταπέσει, 24, 55. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται 24, 56, ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται 24, 57, ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται 2458 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται 24-59 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται 24-60 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται 24-61 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται 2462. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται 2356. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται 2357. 58 που είναι Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται 2463. Ψηφίζουμε. Πέρας. απορρίπτεται 24-64. ψηφίζουμε πέρας κύριος Βίλενη νομίζω ότι μάλλον δεν πιστεύει ότι θα έπρεπε να διακόψουμε για τουλάχιστον ένα τρίλεπτο ναι αλλά μην μου το λέτε στη μέση ψηφοφορίας ψηφοφορίας Ψηφίζουμε την 2464. 2464. Παναλαμβάνουμε τη ζωοφορία. 2464. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Ε, έμεναν λίγες τροπολογίες και έλεγα να τις τελειώσουμε. Αυτή είναι η πρόθεσή μου, γιατί πηγαίναμε γρήγορα, οπότε δεν ήθελα να διακόψω. Περνάμε στην προφορική 9, υπάρχουν στάσεις, υπάρχουν, αλλά δεν ξεχνάμε, προφορική 10, υπάρχουν ενστάσεις. πέντε. πέρας απορρίπτεται 2466 πέρας απορρίπτεται 2467 ψηφίζουμε πέρας απορρίπτεται 2468 και 2397 που είναι ταυτόσιμες ψηφίζουμε πέρας Απορρίπτονται. 2469. Ψηφίζουμε. Πέρασε. 2470. Προηγούμενη απορρίφθηκε. Πέρασε. Απορρίπτεται. 2398 και ένβη 177. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. 2471. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται 2472, 2400 και 2401 και 24... που είναι ταυτόσιμες, ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτονται 2473. Πέρας. Απορρίπτεται προφορική 11. Υπάρχουν στάσεις 2403 ψηφίζουμε. 20 και 04, 24, 04, 24, 03. Ψηφίζουμε, πέρας. Απορρίπτονται. 24.05 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτονται. 24.06 και 07 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτονται. Ε, ε απασχόλησης 85 Ψηφίζουμε πέρας. Απορρίπτεται. 86 της Επιτροπής Απασχόλησης ε, πέρας. Απορρίπτεται. 87 της Επιτροπής Απασχόλησης ε, πέρας. Απορρίπτεται. Και τώρα περνάμε στην 2004. και στις ε, Συγγνώμη, αλλά χάσαμε τα νούμερα που ανέφερε ο Πρόεδρο. 24-13 απορρίπτε. Ε, ξεκινάει. Ψηφοφορία. Πέρα. 24 75 24-55, 24-14 και 24-15. Ταυτόσιμε ψηφίζουμε. Πέρα. Απορρίπτεται. 24-21 ψηφίζουμε. Πέρας απορρίπτεται 24-22 πέρας δεκτή 24-12 22 συγγνώμη 24-24 ψηφίζουμε πέρας απορρίπτεται 2-4-25 ψηφίζουμε πέρας Απορρίπτεται. 2, 4, 26. ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. 24, 27, 28 και 29 Ταυτόσιμες. ψηφιζουμε Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτονται. 24-30 ταυτόσημη με την ΕΒ 178 ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνονται. 24-32 ψηφίζουμε. Mm -hmm. Πέρας. Απορρίπτεται. 24-31 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Τελειώσαμε με τα άρθρα. Ευχαριστώ για τη συνεργασία σας. Λιγότερο από δύο ώρες μας χρειάστηκαν διακόψουμε για 5-6 λεπτά, αλλά ας μην καθυστερήσουμε. Λοιπόν, 5 λεπτάκια και επανερχόμαστε. Vamos. Sí, dime, dime. Vamos entrando. Please. Take your seats. ready to continue. Yeah. Or not? του Τι Okay, Antinoro. I think we are all together again. Bien, una, antes, de, antes de empezar con los Προτού να περάσουμε στα παραρτήματα, θα ήθελα να σας πω, όπως ε, και στα γραπτά, θα δείτε ότι δεν ε, υπάρχουν πολλά λάθη. Ε, Υπάρχουν κάποιε τροπολογίε οι οποίε ε, έχουν καταπέσει και τι ψηφίσαμε. Απλά σα το λέω για να το γνωρίζετε. Αυτό είναι ο απολογισμό λοιπόν των ε, ψηφοφοριών και θα συνεχίσουμε. Έχουν πολλές ε, ψηφοφορίες ακόμα, αλλά θα πρέπει και εδώ να βιαστούμε και θα μπορούσαμε να το πετύχουμε αν αρκεί μάλλον να προσέχουμε. Ξεκινάμε με τα παραρτήματα προπολογια 2436, 2437. Ξεκινάμε. Πέρασε. Εγκρίθηκαν. 2438 ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. 155. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Δεκτή. ψηφίζουμε. Πέρας. δεκτη 2440 ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. Ε, ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 156 ψηφίζουμε. Πέρασε. Δεκτή. Ένβη 179. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Δεκτή. 2.442. Υπέρ. Ε, συγγνώμη. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Δεκτή. 24.43. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. 24-44 ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. 45 ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. Περνάμε τώρα στα εκτιμώντα. Ρέχει 1, 158 και 159 που είναι ταυτόσιμε. Ψηφίζουμε. Πέρασε δεκτές 160 όχι καταπίπτει Okay. No, vamos a la 160. 161. 161 προπολογία ελπίζουμε. 161. Στα εκτιμώντα σελίδα 240. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Sí, está ok, no había ningún. Entonces, volvemos a donde estábamos. 1, 6. 161. 234 σελίδα. Έχεις κάποιο πρόβλημα, Ραούλ? Σελίδα 234 στο ισπανικό προφανώς έγραφο, 2.40 στο ελληνικό. Έχουμε κάποιο πρόβλημα με τη φωτοτυπία, παρατηρεί ο Ραούλ. 1.61, Ζωάο Φερέιρα, ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. Ένβη 1, ψηφίζουμε. Πέρας δεκτή. Ένα του εισηγητή και ρέγγι 2. Ψηφίζουμε, πέρας. Δεκτή, δεκτές. Της απασχόλησης 2 καταπίπτει, περνάμε στην 164. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. Ρέτζι 3. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. Έμπλη 3. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 165. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. Όχι. Έμπλ 4. Έμπλ 4. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 167 ψηφίζουμε. Πέρασε. Δεκτή. Έμπλ 5, 6. Έμπλ 6 ψηφίζουμε. Πέρασε. Δεκτή. Έμπλ 5. 7 ε, συγγνώμη, 7. Πέρασε. Δεκτή. 70. 170. Ψηφίζουμε. Πέρας. Συγγνώμη. Έχουμε κάποιο πρόβλημα με τις φωτολυπίες. Ε, έχουμε χάσει μια σελίδα. Μας έχει ξεφύγει. Ε. Μπορώ να σου δώσω τα δικά μου αν θες, Ραούλ. Ευχαριστώ για την προσφορά, Πρόεδρε, αλλά τα καταφέραμε. 170 πατράω. 170. Ψηφίζουμε. 170. Πέρασε. Δεκτή. 100. Όχι. 172. 172 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 173. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 174. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Δεκτή. 175. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Δεκτή. Εκατόν Ξεκινάμε την ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. 180 ψηφίζουμε πέρας απορρίπτεται 181 ψηφίζουμε πέρας δεκτή Εκατόν ενενήντα ένα.

Προπολογισμό 6. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 7 του προπολογισμού. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 196. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. Έμπλ 10. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 198. Σφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 199. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. Περνάμε στην 200. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 201. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 204. Πέρας. Δεκτή. Περνάμε στην ΕΜΠΛ 12. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 207. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. ΕΜΠΛ 13. Ε, ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 208. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Έμπλου 14. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεχτή. 209. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεχτή. 210. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 213. Πέρας. Δεκτή. 200... 216. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 217. Πέρας. Δεκτή. 200. Όχι. Έμπλ 17. Ψηφίσμα. Πέρας. Δεκτή. 221. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 226. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 227. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. Έπλου 19. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. προπολογία 8. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 228. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 229. Πέρας. Απορρίπτεται. 230. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 231. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Έμπλ 20. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 9 τροπολογία. Φράγει 9. Πέρας. Δεκτή. 232. Πέρας. Δεκτή. 233. Ψηφίζουμε. Πέρας δεκτή. 200, 238. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 239. Πέρας. Δεκτή. 200. Κάνουμε ένα άλμα. Έμπλη 23 με επικοντό ήταν αυτό. Όχι, 248, συγγνώμη. 248. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. Έμπλ 23. Πέρας. Δεκτή. 249. Πέρας Δεκτή 2.58 Ψυχολόγος Πέρας Δεκτή 266 Ψύχισε Πέρας Δεκτή. 13, 267, 268, 69 και 70 που είναι τεπτώσιμες. Ψηφίσουμε. Πέρας. Δεκτές. οκτώ. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 2,79 ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 2,80 και 14 ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτές. τώρα που πάμε. Στη 2, 93, 94, 95, 96, 97 και MV16 ψηφίζουμε. Πέρασε. Δεκτές. Και τώρα Περιμένω τα φώτα σας. Περνάμε στη 16. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτέ. 301. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Δεκτή 302. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. Προεπολογισμός 11. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 12 του προπολογισμού. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 17. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Δεκτή. 17 έγινε δεκτή. 18. Ψηφίζουμε. 18. 18 πέρας της ψηφοφορίας απορρίφθηκε 303 303 ναι. ψηφίζουμε πέρας δεκτή 306 306 Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 307. Πέρας. Δεκτή. Και τώρα φτάνουμε στην 309, 309. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 310, 310. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 3-11. Πέρας. Απορρίπτεται. 3-12. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 3-2-4. Όχι, 3-23. 3-23. Ψηφίζουμε. Δεκτή. Πέρας. Δεκτή. 324. Πέρας. Δεκτή. 23. 23. Προπολογία. Πέρας. Δεκτή. Δεκτή 23. 3-29. 29. Πέρας. Απορρίπτεται. Ένβη 21. Πέρας. Δεκτή. 24. Πέρας. Δεκτή. 330. Πέρας απορρίπτεται 431 ψηφίζουμε λήξη δεκτή 3.32 ψηφίζουμε πέρας δεκτή 3.34 ψηφίζουμε Λήξη ψηφοφορια Δεκτή. 3.35. Ψηφίζουμε. Έληξη ψηφοφορία. Δεκτή. 3.42. Ψηφίζουμε. Έληξε. Δεκτή. 3.48. 3.48 ψηφίζουμε. Έληξη ψηφοφορία. Δεκτή. 3.50. 350. Ψηφίζουμε. Έληξε. Δεκτή. 3.58. Έληξε η ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. 3.59. Ψηφίζουμε. Έληξε. Δεκτή. 3.63. Ψηφίζουμε. Έληξε η ψηφοφορία. Δεκτή. 3.64. <coughs> Δεκτή. 369. Ψηφίζουμε. Έληξε ψηφοφορία. Δεκτή. 370. Ψηφίζουμε. Έληξε. Δεκτή 71, 73, 71, 72 και MV29 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίφθηκε. 373 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίφθηκε. 374 ψηφίζουμε. Λήξεις. Δεκτή. Ρέτζι 20. Συγγνώμη, 3,75. 3,75. Ψηφίζουμε. Λήξεις. Απορρίφθηκε. 3,76. Ψηφίζουμε. Λήξεις. Δεκτή. 3.78. ψηφίζουμε έληξε δεκτή περνάμε στην ε, Apple 31 ψηφίζουμε πέρας δεκτή τροπολογία 382 ψηφίζουμε Πέρας. Δεκτή. 27. Συγγνώμη. Έμπλ 33. 33. Έμπλ 33. Λέξεις απορρίφθηκε. 28 τροπολογία. ψηφίσουμε, Πέρας. Δεκτή. 383 προπολογία. Έληξε. Απορριφθήκε. 384. Ψηφίζουμε. Έληξε. Δεκτή. 391. 391. Ψηφίζουμε. Έληξε. Απορρίφθηκε. 400 τροπολογία. 400. Έληξε την ψηφοφορία. Δεκτή. 402. 402. Τροπολογία. Έληξε. Δεκτή. Τροπολογία 31. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 406, 406 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται 407. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίφθηκε. 32. Τροπολογία 32. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 408. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 410. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Ρέτζι 27. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. Προπολογία 411. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Ρέτζι 28. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 412. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 413. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. Ρέτζι 29. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. NV33. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 416. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 417. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 422. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 423. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 428. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. NV36. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. NV37. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται 430, 430. Πέρας. Εγκρίνεται MV38. Ψηφίζουμε. Έλλειψη ψηφοφορία. Εγκρίνεται 431. Πέρας. εγκρίνεται 432 ψηφίζουμε πέρας δεκτή 433 ψηφίζουμε πέρας απορρίφθηκε 434 ψηφίζουμε πέρας δεκτή Έμπλ 37 ψηφίζουμε πέρας δεκτή 4.35 ψηφίζουμε πέρας απορρίπτεται 4.36 ψηφίζουμε πέρας απορρίπτεται 4.37 ψηφίζουμε Πέρας. Απορρίπτεται. 36 ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 4.38 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 4.39 ψηφίζουμε. Πέρας απορρίπτεται 440 ψηφίζουμε πέρας απορρίπτεται NV40 ψηφίζουμε πέρας δεκτή 441 ψηφίζουμε πέρας δεκτή 451 Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 4.52. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 4.53. Ψηφίζουμε. Πέρας. 141. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτεί. 4.54. Όχι. 4.55. 4.55. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτεί. 4.57. Πέρας. Απορρίπτεται. 4.58 πέρας απορρίπτεται 4.56 ψηφίζουμε πέρας απορρίπτεται έμφυ 42 ψηφίζουμε πέρας Δεκτή. 4.59. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 4.60. Πέρας. Δεκτή. Όχι, απορρίπτεται, συγγνώμη, συγγνώμη, απορρίπτεται. Απορρίφθηκε η 460. Περνάμε στην ε, budget 1, προβλόσμος 1. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 2 του προπολογισμού. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Τρία του προπολογισμού. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. Έχει συμπεριληφθεί και στην τοπολογία 25. Το προπολογισμό 4 ψηφίζουμε. Πέρα. Απορρίπτεται. Και η τροπολογία 157 ψηφίζουμε. Πέρα. Απορρίπτεται. Ο κύριο Καντέκα έχει το λόγο. Τελειώσαμε τι ψηφορίε του πρώτου τμήματο. Σα ευχαριστώ. Δίνω... Τώρα μπορούμε να κάνουμε ένα διάλειμμα 10 λεπτών. Ένα 10 λεπτό λοιπόν διάλειμμα. Ή όχι 5, 5 λεπτών. 5 γιατί έτσι και θα γίνουν 10. Και θα έρθουμε εδώ με την, με την τροπημένη έκθεση και το Δεν νομίζω ότι χρειάζεται ένα διάλειμμα. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο είναι απαραίτητο. Este planteamiento, señor lo habíamos hecho al principio. Κοιτάξτε, αυτό το συμφωνήσαμε άμα την ενάρξη τη συνεδρίαση το πρωί και βεστώσει δεν πρόκειται να χάσουμε και πολύ χρόνο. Γρήγοροι θα είμαστε. Τι έγινε, να μην κάνουμε διάλειμμα, να μην κάνουμε διακοπή. Ε, θα συνεχίσουμε τότε έτσι. Εντάξει, εγώ δεν έχω αντίρρηση. Κοιτάξτε, μισό λεπτό, μισό λεπτό ησυχία στην αίθουσα είχαμε συμφωνήσει να κάνουμε μια διακοπή. Άρα θα έπρεπε να διατηρήσουμε την ε, αρχική μας απόφαση. Κάνουμε λοιπόν ένα πεντάλεπτο διάλειμμα, να ξεμουδιάσουμε και θα επανέλθουμε.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 Ready? Bien, pues están preparados. Vamos a... Είστε πανέτοιμοι λοιπόν να ψηφίσουμε το ψήφισμα νομοθετική πρόταση που οπτροποίηθηκε. Αρχίζουμε η ψηφοφορία. Σέρα. Έληξε. Se πρόβλημα να... Εγκρίθηκε το ψήφισμα χοντικού περιεχομένου ε, και τώρα στο σύνολό τη όπως τροποποιήθηκε η πρόταση ψηφίζουμε. Θύρα. Έληξε ψηφοφορία. Δεκτό. Και τώρα ψηφίζουμε την εντολή για το τριμερή διάλογο όπως ε, ήδη τον ε, γνωρίζετε, το έχετε υπόψη σας. Σιέρα. Πέρα στις Απορρίπτεται. Λοιπόν. Ευχαριστώ ε, όλες και όλους που φροντίσατε να φέρουμε σε αίσιο πέρας ε, τις εργασίες μας ε, και συγγνώμη για τα ενδεχόμενα λάθη τα οποία διέπραξα ως πρόεδρος. Δεν έχουμε τελειώσει όμως. Μας μένουν ακόμα δύο ψηφοφορίε, ε, σύντομες. Παρακαλώ, παρακαλώ. Κύριος Κάντεκ, έχει το λόγο. Παρακαλώ κύριε Κάντεκ, έχετε το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή είμαι η εισηγητής ε, για το θέμα αυτό τον, ε, του Δραμείου ε, Αλληλείας και Θαλασσίων Θεμάτων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις εισηγητές που δούλεψαν μαζί μου για αυτό το, την τεράστια έκθεση. Με τη βοήθειά τους τα κατάφερα όπως επίσης και με την αίσθηση ευθύνης που επέδειξαν όλοι. Σας ευχαριστώ για αυτήν ε, τη θετική ψηφοφορία. Το μόνο που με στεναχωρεί είναι το θέμα της εντολής, γιατί είχα ζητήσει εντολή, αλλά τέλος πάντων εντάξει. Καθυστερεί απλώς λίγο περισσότερο τις συζητήσεις, αλλά δεν είναι ε, πολύ σοβαρό, γιατί ούτως ή άλλως θα ψηφίσουμε και στην Ολομέλεια και μετά από την Ολομέλεια θα αρχίσουμε τον τριμερή διάλογο με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Θα μπορούσαμε να είχαμε ξεκινήσει λίγο πιο νωρί, αλλά τέλο πάντων δεν πειράζει, θα αρχίσουμε λίγο παραπάνω. Σα ευχαριστώ πάντω για όλα. Ευχαριστώ κύριε Καντέκ. Περνάμε στο επόμενο σημείο τη μέσης διατάξεω, εντάχει. Πρόκειται για την ε, ψήφιση τη έκθεση του κυρίου Νικουλέσκου το υπαριθμό 6 θέμα στην μεσοδιάταξη. Σχετικά με τη διατήρηση των ελευθερικών πόρων ε, μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλασσίων οργανισμών ή γόνων. Περνάμε λοιπόν στη ψηφοφορία, στην τροπολογία 2. Έληξε ψηφοφορία, ησυχία παρακαλώ και ηρεμία ζητώ. Δεκτή. Τροπολογία υπερθυμών 5. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία υπερθυμών 10. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία υπερθυμών 6. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 7. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 8. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία υπαριθμών 1. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία υπαριθμών 9. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. Ψηφίζουμε τώρα την τροποποιημένη νομοθετική πρόταση πέρα ψηφοφορία. Δεκτή. Και τώρα το ψήφισμα νομοθετικού περιεχομένου. Ψηφίζουμε πέρας. Δεκτό. Συγχαρητήρια κύριε Νικουλέσκου. Περνάμε στο επόμενο σημείο, σημείο 7 τη μης διατάξεω, ε, ιδιωτικά με τη διατήρηση των δευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων στα ύδατα τη Βαλτική θάλασσα τον Beltke του Sound, έκθεση του κυρίου Βαλέσα. Προπολογή παθμό 5. Ψηφίζουμε, πέρας. Απορρίπτεται 6. Προπολογία ψηφίζουμε, πέρα Απορρίπτεται. Προπολογία 7. Ψηφίζουμε. πέρα. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 2. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 3. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. Η 4 έχει καταπέσει. Ψηφίζουμε τώρα την προηγουμένη πρόταση πέρα ψηφοφορίας νεκτή και τώρα το ψήφισμα νοχωρικού περιεχομένου πέρας δεκτό Συγχαρητήρια κύριε Βαλέσσα και σας ευχαριστώ όλες και όλους αυτό επίση και τι υπηρεσίε. ο πρόεδρος ευχαριστεί τους και οι Γερμηνείς ευχαριστούν τον πρόεδρο. Ah, Κοιτάξτε, υπάρχει ένα εκρεμέ ζήτημα που μου θύμισε ο φίλος και συνάδελφος ε, στην μέσα διάταξη δεν ε, εγκρίναμε την μέσα διάταξη πρώτα απ' όλα. Το σημείο 2. Δηλαδή αυτό που αναφέρεται στην έγκριση της ημερησίας διατάξεως. Ε, το ξεχάσαμε. Η συνάντηση με την κυρία Δαμανάκη θα γίνει και κλεισμένο των θυρών. Εντάξει, ξεχάσαμε να εγκρίνουμε την διάταξη, δεν νομίζω